Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτές τις ερωτήσεις για τον εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων κατόπιν ετοίματος Πρόεδρου της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τον ανταγωνισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την παρουσία της Κομισιόν για να ποντήσει και λυπάμαι που δεν μπόρεσε να είναι επίτροπος αντιπρόεδρος Αλμούνιας καθώς ε, είναι υπεύθυνο ε, της ναι. πολιτικής ανταγωνισμού. Η πρωτοβουλία για τον εξεχρονισμό των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων που ξεκίνησε από την Κομισιόν πέρσι το Μάιο και είναι η αιτία των δύο προτάσεων ε, κανονισμού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων μαζί με τις υπόλοιπες πτυχές της πολιτικής ανταγωνισμού αποτελεί ένα θεμελιώδες μέρος του σχεδίου της ενιαίας αγοράς. Οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να συνεισφέρουν στο να διορθώσουν τα κενά της αγοράς και να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον χωρίς να βλάψουν την οικονομία στο σύνολό τους ούτε να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην αγορά υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις που παράγουν αγαθά ή παρέχουν επιχειρήσεις ε, των οποίων η παροχή δεν μπορούσε να γίνει με άλλο τρόπο. Σε δύσκολους καιρούς, ε, στο πλαίσιο ε, της εποχής δημοσιονομικής εξυγίανσης και αδύναμων οικονομιών, είναι περισσότερο επιτεκτικό από ποτέ να έχουμε αποτελεσματικές δημοσίες δαπάνες και ε, μπορεί να έχουν δημόσιες δαπάνες καλύτερο αντίκτυπο να έχουμε ένα αφιές σύστημα κρατικών ενισχύσεων που επιστηρίζουν τα δικαιώματα των αφορολογουμένων και των ανταγωνιζόμενων και που να αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο μέγιστης ασφάλειας δικαίου με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία. Η Επιτροπή βεβαιώνει όταν ε, θα προωθήσει μία αναθεώρηση για να εφαρμοστούν σωστά οι κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, επικεντρωνόμενοι στα μέτρα που μπορεί να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό με μεγαλύτερη αυστηρότητα, χωρίς να δημιουργούνται μία απαραίτητα εμπόδια για τα μέτρα που έχουν επιπτώσει στο διασυνοριακό εμπόριο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη στόχων όπως οι περιφερειακές επενδύσεις, η έρευνα και η ανάπτυξη, η προώθηση του πολιτισμού, μεταξύ άλλων. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να προωθηθούν, αλλά δεν είναι καινούργοι, γιατί επιδιώχθησαν και από άλλους ηθήνοντες της πολιτικής ανταγωνισμού. Γι' αυτό, καθώς ε, πρόκειται για την πρώτη ολομέλεια, φέτος ε, θέλω να στείλω τις καλύτερες ευχές μου για να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία από τους προκατόχους σας. Γι' αυτό πρέπει να τελειοποιηθεί το σύστημα. Το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για τις κρατικές ενισχύσεις που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2011 πρότεινε ήδη την αναγκαιότητα βελτίωσης του ελέγχου των εθνικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή ε, εντόπισε ότι στο 40% των περιπτώσεων που ελέγχονται για τα μέτρα εξαίρεση σε μπλοκ που υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζουν πρόβλημα. Θα ε, χρειαστεί λοιπόν να ληφθεί δράση σε διάφορες κατευθύνσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη διαβούλευση εκ των προτέρων, βελτιώνοντας το συντονισμό έτσι ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται συνεκτικά, βελτιώνοντας ε, τη συμμόρφωση με τα μέτρα που έχουν θετηθεί σε εθνικό επίπεδο και με το να γίνεται μια πλήρης παρακολούθηση με τη διάθεση και των κατάλληλων πληροφοριών που σχετίζονται με την ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων. Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων έχει μεγάλη οικονομική και πολιτική σημασία. Θυγεί αποφάσεις που έχουν εθετηθεί από αρχές εθνικό επίπεδο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά η άσκηση αυτών των εξουσιών και ο έλεγχο τη στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τμήμα τη δημοκρατική λειτουργία τη Ένωση. Πέραν αυτού, οι νέε προτάσει ε, προετοιμάστηκαν βάσει του άρθρου 109 τη Συνθήκη τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναγνωρίζει στο Κοινοβούλιο έναν απλά ε, συμβουλευτικό χαρακτήρα. Άλλε πτυχέ τη οικονομική διακυβέρνηση ήδη ήταν αντικείμενο συναπόφαση όπως και μία από τις προτάσεις που τέθηκαν, που τροποποιεί ένα μέσο που εθετήθηκε προηγουμένως μέσα στην απόφαση σε σχέση με τις υποχρεώσεις της, ε, των δημοσίων υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών. Δεν πρέπει να ξεχνάει η Κομισιόν ότι το Κοινοβούλιο είναι η πηγή της νομιμότητάς του και πρώτος συμμαχός της. Θα ήθελα η Κομισιόν να επιβεβαιώσει τα δύο ακόλουθα ζητήματα. Καταρχήν, αν θα λάβει υπόψη τη γνωμοδοτήση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τι αναφερόμενε προτάσει και δεύτερον, στο πλαίσιο μια μελλοντική τροποποίηση τη συνθήκη θα συμφωνούσε ότι η έλλειψη διαδικασία στην απόφαση λόγω τομέα θα πρέπει να θεωρηθεί με σκοπό να υπάρξει ευθυγράμμιση αυτού του τομέα με άλλε πτυχέ που αφορούν τι οικονομικέ ρυθμίσει. Ευχαριστούμε κύριε Πρεσέντο. Και τώρα εκ μέρους της Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος Κάλλας. Κυρία Κυρίες και κύριοι, η Κομισιόν χαιρετίζει το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα του εξυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων και έχει ήδη υποβάλει σχετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου του 12. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον διάλογο που υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων. Η προσφορά του Κοινοβουλίου, οι προτάσεις του που άρχισαν από την εικόνα το Σεπτέμβριο του 12 ως σχόλιο του προγράμματος δράσεις της Επιτροπής ήταν και αυτές πολύτιμες για μας. Οι δύο προτάσεις μας ε, υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη ταυτόχρονα μετά την έγκρισή του την 5η Δεκεμβρίου όπως σας είπα προηγούμενες διαβουλεύσεις για τις κύριες κατευθύνσεις των προτάσεων αυτών υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο εκ των προτέρων όπως και στα κράτη-μέλη. Με βάση το άρθρο 109 της Νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαβούλευση του Κοινοβουλίου με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Κομισιόν σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο θέλει να συμπεριληφθεί μια διαδικασία συναπόφασης για αυτά τα θέματα σε πιθανή αναθεώρηση των συνθήκων. Αλλά αυτό ξεπερνάει το νομικό πλαίσιο επί του οποίου βασίζονται αυτές οι, οι δύο προτάσεις που συζητούμε. Η Κομισιόν είναι αποφασισμένη να κρατήσει, να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο για κάθε τέτοια πρωτοβουλία και τέτοιες καινούργιες διαβουλεύσεις και προσβλέπει στον ορισμό των εισηγητών για τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για τις δύο αυτές προτάσεις. Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες για τους εισηγητές αυτούς και άλλους ενδιαφερόμενους ευρωβουλευτάς για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων και για οποιαδήποτε αποσαφήνιση. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα εξ ονόματος του ΕΛΚ, κύριε Χόκμαρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τον Επιτροπό. Πρέπει να θυμόμαστε πως οι κρατικές ενισχύσεις πάντα αποτελούν κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού και ε, βεβαίως πάντα υπάρχει κίνδυνος διατήρησης παλαιών δομών εις βάρος των νέων ε, νέων εισερχόμενων και των νέων ιδεών. Γι' αυτό έχουμε νομοθεσία περί ανταγωνισμού και αυστηρούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Και όταν μιλάμε για εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων, νομίζω πως πρέπει να βάλουμε στην κατεύθυνση λιγότερων αλλά πιο στοχευμένων κρατικών ενισχύσεων. Μόλις έγινε η συζήτηση για τα δημόσια οικονομικά. Και βεβαίω οι κρατικές ενισχύσει πάντα υπονομεύουν τη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών. Γι' αυτό ο στόχο πρέπει να είναι λιγότερε και πιο στοχευμένε κρατικές ενισχύσει να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη γνώση τη δέσμε καινοτομία, αλλά όχι να στηρίζουμε διαφορετικές εταιρείε, να υποστηρίζουμε την ανάδυση νέων τεχνολογιών σε διάφορους τομείς και νομίζω πως επαφείται στην Κομισιόν να φροντίσει να υπάρξει μια συνέχεια, να έχουμε λιγότερες κρατικές ενισχύσεις για να δώσουμε την δυνατότητα να έχουμε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και περισσότερο ανταγωνισμό και όπως είπα να μην έχουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού αλλά να βοηθήσουμε στην περισσότερη καινοτομία και νέες υποδομές και πόλους επιστήμης. Σας ευχαριστώ κύριε Χέκμαρκ, ο κύριος Κοφεράτη για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, φαντάζομαι ότι και εσείς όπως και εμείς θέλετε να εργάζεστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα ήταν απαραίτητες πλέον οι κρατικές ενισχύσεις. Όμως αυτό είναι ιδανικό πολύ μακρινό. Σήμερα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι απαιτήσει συναρμόνιση των παραγωγικών τομέων και των διάφορων οικονομικών διαστάσεων είναι δυνατό μόνο αν η πολιτική αυτή παραμείνει. Και επίσης είναι αλήθες ότι αν όπως σήμερα φτάσουμε σε τόσο δύσκολες καταστάσεις επειδή η κρίση χτυπά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ο κίνδυνος, οι κρατικές ενισχύσεις να καταστούν ε, και μια υπερβολή αυτονομίας ε, χρήσης ε, της να γίνουν μία από τις συνθήκες που τροποποιούν τον ανταγωνισμό και ε, τη δυναμική των οικονομικών σχέσεων. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικός ο εξυγχρονισμός, πρέπει να στραφούμε προς αυτόν, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει. Νομίζω ότι υπάρχει ένα προφανές πρόβλημα χρόνου. Αν υπόκειται σε ιδιαίτερα μακρές διαδικασίες κρατικές ενισχύσεις όπως σήμερα, μπορεί να μην έχουν την απαραίτητη αποτελεσματικότητα για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις κρίσης που μπορεί μάλιστα να γίνουν πραγματικές ε, καταστάσεις ανάγκης. Δεύτερον, αν χρειάζεται ένας έλεγχος ε, του τρόπου ε, που χορηγούνται οι κρατικές ενισχύσεις για να αποφευθεί η κατάχρηση και για να αποφευθεί οι κρατικές ενισχύσεις να διοχετευτούν προς κάποιους δικαιούχους διαφορετικούς από αυτούς που είχαν δηλαδή στην αρχή. Πρέπει λοιπόν να βιαστούμε και πρέπει να υπάρχει όμως και ένα συνεχής έλεγχος και θα είναι πιο έλεγχο να υπάρχει αυτός ο έλεγχος αν η διαδικασία, όπως λέει και η Κομισιόν, καθοριστεί σύμφωνα με παραμέτρους και κριτήρια που θα πρέπει να επιβεβαιώνονται όχι μόνο από την πρακτική και την εμπειρία, αλλά και από κάποια καινοτόμα στοιχεία. Ένα τρίτο στοιχείο σε ό,τι αφορά τον εξεχρονισμό ε, είναι η σχέση μεταξύ των διαφόρων θεσμικών επιπέδων Συμβουλίου, Κομισιών Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να έχει ένα ρόλο στο περιθώριο. Η μόνη διαβούλευση του Κοινοβουλίου και εγώ ε, λαμβάνω υπόψη αυτό που είπατε εδώ, ότι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη η άποψη του Κοινοβουλίου και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, αλλά αν αυτό το δεν ε, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο ζήτημα, δεν θα κάνουμε ένα βήμα πραγματικά προς τα μπρος. Εμείς ε, σας ζητάμε ένα βήμα για το μέλλον, γιατί γνωρίζουμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι συνθήκες. Πρέπει στο μέλλον να προβλεφθεί ένας πρωταρχικός ρόλος για το Κοινοβούλιο και όχι απλώς ένας ρόλος απλής εμπλοκής. Ευχαριστούμε κύριε Κοφεράτη και τώρα εκ μέρους των φιλελευθέρων Σοφίντφιλτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Αισθάνομαι κάποια ανησυχία διαβάζοντας ε, την πρόταση. Κάποια τα στοιχεία έχουν ήδη αναφερθεί από τους συναδέλφους, ειδικά ε, τον ε, κύριο Σαντισφρεσέδο και τον κύριο Χέκ γιατί ο στόχος ακούγεται υπέροχος, λιγότερη και πιο στοχευμέ... λιγότερες και πιο στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις. Τα ακούμε εδώ και χρόνια, αλλά έχω την αίσθηση πως οι προτάσεις αυτές βασικά στόχο έχουν αφενός να γίνει πιο εύκολο να δοθούν κρατικές ενισχύσεις και να γίνει πιο δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς αυτές τις ενισχύσεις. Για εταιρείε παραδείγματο χάρη που θεωρούν πως έχουν έτσι ένα μειονέκτημα ε, οι κρατικές ενισχύσεις υποτίθεται πως είναι κάτι το εξαιρετικό και το προσωρινό. Ο κύριος Κοφεράτη μόλις ανέφερε ε, πως ε, σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους πρέπει να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης, αλλά έχω την αίσθηση πως με όλες τις τροποποιήσεις του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων τα τελευταία χρόνια γίνεται κάτι το διαρθρωτικό πλέον, κάτι το, που είναι μέρος των τακτικών δημοσίων δαπανών. Και δεν είναι δυνατόν να είναι αυτό. Το σκεπτικό μας πρέπει να παραμείνει κάτι το εξαιρετικό. Επίσης δεν απαντήθηκε το ερώτημα που σωστά ετέθη ε, από τον κύριο Σάντσες Πρεσέδο για την έκθεση που τονίζει πως πράγματι νομίζω γύρω στο 40% των ενισχύσεων που δίνονται ε, υπό το καθεστώς τη εξαίρεσης ε, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και ίσως είναι τελείως αδικαιολόγητες. Πώς μπορούμε να μιλάμε για χαλάρωση του καθεστώτος κρατικών ισχύσεων αν δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα. Και τέλος, ε, συμφωνώ με όσους είπαν πως τελικά ε, το θέμα δεν είναι απλώς διοικητικό, αφορά πολιτικές επιλογές και νομίζω πως έχει φτάσει η στιγμή η Κομισιόν να συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο. Έχει φτάσει η στιγμή να ε, αποτελέσει και αυτό το ζήτημα αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ κυρία Ινετφέλτ. Τον λόγο έχει ο κύριος Σβάμπ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως συμφωνώ με μέρη με αυτό το οποίο υπόθηκε, αλλά θέλω να πω πω ακόμα και αν δεν είναι εδώ πέρα σήμερα ο κύριος Αλμούνια, οπωσδήποτε η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να ε, επικεντρωθεί στις ε, σημαντικές και δύσκολες περιπτώσεις και βεβαίω επί της αρχής είναι σωστή αυτή η πρόταση επί της αρχής. Πρέπει όμως να δούμε πραγματικά τις σημαντικές περιπτώσεις. Θεωρώ πως τα σημεία στα οποία ασκήθηκε κριτική από τους συναδέλφους όπως από την κυρία Ίνετφελτ πράγματι ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι' αυτό πρέπει η Κομισιόν να αναπτύξει λεπτομερή κριτήρια με βάση τα οποία θα υπάρξει ένας καθορισμός των περιπτώσεων. Δεύτερον, κυρία Πρόεδρε, όσο ε, η, στο μέτρο που η Κομισιόν θέλει να αποσυρθεί από τον εξάντε έλεγχο και να επικεντρωθεί στον έλεγχο εκ των υστέρων, ex θα πρέπει να φροντίσουμε οι εθνικές αρχές να αναλάβουν αυτό το καθήκον και να το εκτελούν με τρόπο συνεπή. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφενός και Εθνικών Αρχών αυτέρου η οποία θα βελτιωθεί. Τρίτον, η Κομισιόν λέει πως θα έρχεται σε άμεση επαφή με τα μέρη εκείνα τα οποία έχουν κάποια καταγγελία, καταγγελία για τις περιπτώσεις και μάλιστα θα περιορίζεται στην ουσία της καταγγελίας. Εγώ δεν ξέρω, γιατί εδώ πέρα μιλάμε βεβαίως για δαπάνη χρόνου και πόρων, το εάν υπάρχει και αν δικαιολογείται αυτή, αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει και αν δικαιολογείται αυτή η δαπάνη. Και βεβαίως ε, ήδη έχει αναφερθεί πως ε, τα δίκτυα ευρυζωνικότητας όσον αφορά τη χρησιμοποίηση για λόγους υγείας εξαιρούνται, οπότε υπάρχει ήδη ένας τρόπος για να ε, δείξουν κάποια ελαστικότητα ή οτά και να ξεφύγουν από το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σας ευχαριστώ κύριε Σφάμπ. Περνάμε στην συνάδελφο Γκάλ Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ πως οι κρατικές ενισχύσεις και ο έλεγχο τους πρέπει να βελτιωθούν, να βελτιωθεί η εποπτεία της ε, Κομισιόν για να μην έχουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ο δε σχετικός κανονισμός είναι εξόχως περίπλοκος ε, και αυτό καθιστά και είναι ο ίδιος για μεγάλες και μικρές περιπτώσεις και αυτό επίσης ε, οδηγεί σε περιπλοκότητα. Θεωρώ πως ε, λογικό θα ήταν να ασκεί και εδώ πέρα δημοκρατικό έλεγχο το Κοινοβούλιο. Γιατί δεν υπάρχει εδώ συναπόφαση. Πρέπει να συνεννοηθούμε και να υπάρξει και ένας συντονισμός με τον ε, τομέα με τους τομείς υπόλοιπους της οικονομικής πολιτικής και ο δες έλεγχος ex post δεν επαρκεί. Αν θέλουμε να μιλάμε για πολιτική ανάπτυξης και αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει και συναπόφαση κοινοβουλίου. <clears throat> για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο, η συνθήκη μάλλον λέει ότι κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων που είναι συμβατές με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μπορούν να αποφασιστούν από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Κομισιόν τον Μάιο του 12 η Κομισιόν έκανε προτάσεις για τον εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων και δήλωσε ότι θα κάνει διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και άλλους ενδιαφερόμενους για την εξυγχρονισμό ακριβώς αυτών των κρατικών ενισχύσεων. Η τροπο... Οποιαδήποτε τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να γίνει με διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Εάν η Κομισιόν αποφασίσει να παρατείνει το εύρος αυτών των κανόνων ή να χορηγήσει εξαιρέσεις τότε τα κράτη-μέλη θα έχουν την υποχρέωση να χορηγήσουν, να εφαρμόσουν σωστά τους νέους κανόνες και η διαδικασία θα απλοποιηθεί. Ευχαριστώ. vážená pani predsedajúca vážený pán komisár je pochýb o tom že právne normy je vhodné v prípade Αναμφισβήτητα, η νομοθεσία πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της καθημερινής ζωής από τη σκοπιά αυτή η πρωτοβουλία της Κομισιόν να Υιοθετήσει δύο κανονισμούς για τον ξεχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων. Όμως είναι το, υπάρχει το θέμα της νομικής βάσης. Η Κομισιόν δεν έλαβε υπόψη το, νομικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υπάρχει η απόφαση που θίγει ε, τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέκεται ε, στην κατάρτιση της πρότασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 209 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, φαίνεται λάθος ο τρόπος που προχώρησε η Κομισιόν και ε, το Κοινοβουλίο προτείνει να υπάρξει συναπόφαση στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ο εξυγχρονισμός δηλαδή των κρατικών ενισχύσεων. Μιλάμε εδώ πέρα για ενισχύσεις, οι οποίες στηρίζουν επενδύσεις των εταιριών και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποκτήσει ένα λόγο σε αυτό το ζήτημα, στον ε, εξυγχρονισμό των ε, ενισχύσεων και την αλλαγή του κανονισμού. Δυστυχώς ε, το Κοινοβούλιο έχει μόνο δικαίωμα διαβούλευσης παρά το ότι όπως είπα ο μηχανισμός αυτός έχει σημαντική πολιτική λειτουργία και αποτελέσματα. Η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, δημιουργούνται με τις κρατικές συνεχείς θέσεις εργασίας, ε, βελτιώνεται η οικονομία και υπάρξει και καλύτερη ισορροπία μεταξύ των κλάδων της οικονομίας. Ευχαριστούμε κύριε Μπάνκη. Ο Επίτροπος έχει τώρα τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Οπωσδήποτε τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι συνεχώς στα θέματα τα οποία απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχώς ασχολούμαστε με τις κρατικές ενισχύσεις και ε, ε, με τις προτάσεις ε, κρατικών ισχύσεων και την πιθανή κατάχρησή τους από κράτη-μέλη που θέλουν να ενισχύσουν κάποιες εταιρείες. Ο στόχος μας είναι να το ελέγξουμε αυτό το θέμα. Οπότε είναι ε, αποστολή μας να μην επιτρέψουμε ε, κρατικές ενισχύσεις οι οποίες θα διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Αλλά η ζωή συνεχίζεται, οι καιροί αλλάζουν, οι κανόνες αλλάζουν, η οικονομία αλλάζει και έτσι προσπαθούμε να κάνουμε τους κανόνες αυτούς ε, πιο διαφανείς, ε, κάτι το οποίο έχει κορυφαία σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για την ε, νομική βάση και την οργάνωση αυτού του έργου. Βεβαίως αυτό είναι η απόφαση όλων των νομοθετικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σας διαβεβαίω εξ ονόματος Κομισιόν πως τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς. Σε όλες τις περιπτώσεις ε, και μέσω της διαδικασίας της διαβούλευσης που προβλέπετε στην περίπτωση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ότι έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις επιτρεπόμενες διαστάσεις και το βάρος ορισμένων οδικών οχημάτων. Και θέλω